Ε, για ένα ενιαίο και συνεπέ ευρωπαϊκό πλαίσιο για την εποπτεία τη αγορά. Σα ευχαριστώ ξανά για αυτό, την πολύ καλή, για αυτό το πολύ καλό ψήφισμα. Σα ευχαριστούμε πολύ, κυρία Επίτροπε. Με αυτή την παρέμβαση ολοκληρώνεται η συζήτηση και η ψήφιση των αντίστοιχων προτάσεων ψηφίματο θα γίνει αύριο το μεσημέρι, 12.00. Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη όπου από πλευρά του έχουμε μια κυρία, μια συνάδελφο κυρία, την κυρία Βραζή, που είναι η έκθεση για την διαχείριση της γρήπης ΙΤΑ 1-1. Θα λάβει τον λόγο η συγγήτρια, η κυρία Ριβοζή, για τέσσερα λεπτά. Έχετε τον λόγο, κυρία Ριβοζή, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η γρήπη ΙΤΑ 1-1 είχε πολλές, σημείωσε πολλές απώλειες. Πέρασαν από τότε σχεδόν δύο χρόνια και ο διεθνής Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε κηρύξει έκτακτη κατάσταση επίπεδου 6, το ανώτατο δηλαδή. Πράγμα το οποίο με τη σειρά του οδήγησε την Ευρώπη να λάβει ορισμένα μέτρα όπως καμπάνιες πάρα πολύ ακριβές ε, για εμβόλια, εμβολιασμού και που αποδείχτηκαν τελικά λιγότερο χρήσιμες από ό,τι προέβλεπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σημειώθηκαν 2.900 θάνατοι στην Ευρώπη από τότε, δηλαδή αριθμοί πολύ κατώτεροι από την συνήθη εποχιακή γρήπη, που αριθμοί που υπολογίζονται σε πάνω από 40.000 νεκρούς κάθε χειμώνα. Το δε κόστος ήταν περίπου 1,3 δισεκατομμύρια στο Ηνωμένο Βασίλειο και πάνω από 700 εκατομμύρια στη Γαλλία. Αυτά σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ελεκτικού μας συνεδρίου. Η αξιολόγηση λοιπόν της διαχείρισης της κρίσης αυτής δείχνει ότι υπήρξε δυσανάλογη ανταπόκριση της Ένωσης και των χωρών μελών μεμονωμένα. Προσπαθήσαμε λοιπόν με τους συναδέλφους τους οποίους και ευχαριστώ να καταθέσουμε μια τροπολογία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 εφόσον εγγυάται ο κατασκευαστή την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των εμβολίων του. Τώρα για την ανεξαρτησία, η ταχεία διαδικασία ανάλυσης έδειξε ότι δεν έχουμε τα απαραίτητα επιστημονικά στοιχεία. Οι λύσεις των ιών, οι ιολογικές αναλύσεις πρέπει να γίνονται ανεξάρτητα και διαφανώς καθώς και πλήρως για οποιοδήποτε προϊόν θα χρησιμοποιηθεί σε τέτοιου είδους υγειονομικές επίγουσες ανάγκες. Και την αξιολόγηση, η αξιολόγηση πρέπει να δημοσιεύεται. πάμε ιδιαίτερα γιατί θα ήθελα την αξιολόγηση αυτή να την ελέγχουν και όσοι οργανισμοί προσλαμβάνουν τους εμπειρογνώμονες, αλλά αυτό δεν έγινε δεκτό. Τέλος τονίζω τις περιπτώσεις ναρκοληψίας που σημειώθηκαν στη Σουηδία μετά από τον εμβολιασμό. Καταρχήν, υπάρχουν ακόμη, δείχνει αυτό, σκοτεινές ζώνες ως προς την αποτελεσματικότητα του εμβολίου και μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι που δεν τους έχει λάβει υπόψη ο κατασκευαστής. Η Φιλανδία απαγόρευσε τα εμβόλια αυτά. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία των Φαρμάκων όμως όχι, γιατί περιμένει ακόμη να έχει περισσότερα στοιχεία πριν περιορίσει το εμβόλιο αυτό. Θα ήθελα η Κομισιόν να λάβει τη θέση της Φιλανδίας, γιατί η αρχή της φρόνησης πρέπει να ωφελεί τον ασθενή και όχι μόνο τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστούμε Μισελ. Έχουμε δέκα συναδέλφους που ζητούν να παρέμβουν στη διαδικασία Catch the την ίδια στιγμή, μόλις ολοκληρωθεί το λεπτό, θα φερώ τον λόγο, διότι έχει ο χρόνος προχωρήσει πολύ και πιέζει. Και ο ίδιος ο κανονισμός από την άλλη πλευρά αυτό προβλέπει. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Ντελβό θα λάβει πρώτη τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε έτοιμοι στην Ευρώπη να αντιμετωπίσουμε μια πανδημία. Η απάντηση είναι ναι, αλλά υπάρχει και ένα αλλά με κεφαλαίο α γρήπη H1N1 του 2010 έδειξε ότι το κάθε εθνικό κράτο μέλο ε, λειτουργήσε για λογαριασμό του χωρί μεγάλη αλληλεγγύη και χωρί συνέπειε στι κινήσει. Ω και ο για αυτό το θέμα, πιστεύω ότι έπρεπε να γίνουν αυτέ οι διαπιστώσει. Κυρίω όμω θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε επικοδομητικοί και λίγο πιο συγκεκριμένοι για το καλό των πολιτών μα. Και νομίζω ότι πρέπει να του ε, αποδείξουμε ότι η εμπιστοσύνη που έχουν χάσει σε εμά μπορεί να ανακτηθεί. Ε, πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη αυτέ τι βασικέ προτεραιότητε που μεταξύ άλλων είναι η ενίσχυση τη ε, συστημική συνεργασία μεταξύ κρατομελών, ο καλύτερο συντονισμό με του ευρωπαϊκού φορεί τη υγεία, ε, η διευκρίνηση ε, του ρόλου των ε, φορέων τη Ευρώπη που διαχειρίζονται του υγειονομικού κινδύνου, μια καλύτερη στρατηγική για τα εμβόλια και περισσότερη επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών. Είναι καλή η έκθεση, συγχαίρω την εισηγήτρια για το κείμενο αυτό, αλλά παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να παραμείνει κενό γράμμα. Είναι ευθύνη των κρατών μελών να διατηρήσουν δείξουν ε, και να φέρουν πέρα, να αναλάβουν τις ευθύνες εδώ που έχουν στο θέμα αυτό. Πραγματικές ευθύνες αντί των πολιτών μας. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Ο κύριος Ταμπαζδί παρακαλώ. Muchas gracias. Ο 2009-es influenza világjárvány. Σε ευχαριστώ πολύ. Το κατά το παρελθόν κάποια κράτη-μέλη ήταν τα καλύτερα προετοιμασμένα παγκόσμια εναντί αυτή τη απειλή. Συμφωνώ όμω με του προορίσαντε. Δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ κρατών μερών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακολουθήθηκαν διαφορετικέ πολιτικέ. Σε κάποιε κυβερνήσει από πρώην σοσιαλιστικέ χώρε που ξεκίνησαν καλά σε σχέση με τη γρήπη. Ε, υπήρχε όμως ε, εσωτερική αντιπαράθεση για αυτό το θέμα. Είχαμε κυβερνήσεις που δεν έκαναν τίποτα για την ΙΤΑ ε, 1 Όλα αυτά δεν είναι θετικά. Πρέπει συντονισμένα να δρούμε πάντα. Συμφωνώ απόλυτα ε, με την εισήγηση. Πρέπει να συντονίζουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα εμβόλια. Χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα είναι σωστή η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων. Θέλουμε να γνωρίζουμε όχι μόνο την γεωγραφική διάχυση της γρήπης και των συμβάντων, αλλά θέλουμε να ξέρουμε και τις περιπτώσεις ε, θνησιμότητας ε, για να δρούμε καλύτερα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γιανακουδάκη παρακολουθεί. Uh, thank you. Ευχαριστούμε. Πριν από ένα χρόνο, μια ομάδα βουλευτών συγκεντρωθήκαμε στι Βρυξέλλε για μια τύπη συνάντηση με τον κοινό στόχο να κάνουμε κάτι για τη γρήπη αυτή. Ενώ εξελισσόταν η συνάντηση, ανακάλυψα ότι υπήρχαν τα ίδια εμβόλια, αλλά είχαμε διαφορετικέ προσεγγίσει. Η έκθεση αυτή ήταν μια ευκαιρία το Κοινοβούλιο να αναλάβει θετική δράση ώστε να προετοιμαστούμε για μια μελλοντική πανδημία. Εγώ φοβάμαι ότι εδώ χάθηκε βέβαια μια ευκαιρία. Πολλά σημεία τη έκθεση αυτή είναι αμφισβητήσιμες ε, ε, αξίας, διότι δείχνουν ότι παρόλο που πολλά είναι εφικτά, έχουμε διαφορετική αίσθηση ασφάλειας. Εδώ πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα και να καθορίσουμε μια κοινή προσέγγιση βάσει των όσων μας μάθαμε. Εδώ δεν θέλουμε να επονιδήσουμε κανένα, αλλά αυτό κάνει δυστυχώς η έκθεση, κάτι που θα αποξενώσει πολλούς από του ε, φορεί τη αγορά. Εδώ αυτό ήταν πιο πολιτική σημασία παρά πρακτική. Σε ευχαριστούμε τώρα, κυρία Φιγκερέντο, παρακαλώ. Όχι. Ε, τότε Φερέιρα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε από τα μαθήματα που πρέπει να συναγάγουμε σε σχέση με διαχείριση για την ΙΤΑ 1 τη γρήπη πρέπει να αναγνωρίσουμε την ανάγκη να δημιουργήσουν συστήματα δημόσιας υγείας και προστασίας ε, τα κράτη-μέλη που θα είναι ικανά να δρουν σε ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων. Επίσης ε, διάχυση πληροφοριών για τα φάρμακα που χρειάζονται ιδιαίτερα για ε, μια πανδημία. Η εκπόνηση και αξιολόγηση επιστημονικών μελετών ανεξάρτητων από τη φαρμακοβιομηχανία για την αποτελεσματικότητα και για τη, σχέση ωφέλους ε, και κόστους ε, των φαρμάκων που συνιστούμε. Επίσης, ενίσχυση του δυναμικού για την αντιμετώπιση κινδύνων και στο επίπεδο έρευνα στον τομέα αυτό. Καθώς επίσης και προληπτικά μέτρα για τον τομέα της δημόσιας υγείας. Πρέπει επίσης τέλος να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εθνικών υπηρεσιών και μεταξύ αυτών των θεσμικών διεθνών οργάνων περιφερειακών που έχουν σχέση με αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ κύριε Φερέρα. Λέει ο Πρόεδρος τώρα. Ο κύριος Πάσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφε. Το 2009 ανακάλυψε τα πρώτα κρούσματα γρήπης ε, σε ανθρώπους. Και τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε τα πρώτα προειδοποιητικά μηνύματα. Εκεί επηρεάστηκαν ε, οργανισμοί διεθνούς εμβέλειας όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Παρακολούθηση των Πανδημιών και μάστηκαν πολλά εμβόλια σε μεγάλες ποσότητες ώστε να είναι διαθέσιμα για όλους τους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Εδώ λοιπόν με μετά τι προτροπέ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία και του ΩΣΑ, η Δημοκρατία τη Τσεχία αγόρασε πάνω από 10 δισεκατομμύρια εμβόλια, προκειμένου να είναι προετοιμασμένη για το 2010. Όμω, ε, τελικά δεν πίστεψε κανεί τον ΟΑΣΕ ε, στην περίπτωση αυτή από ό,τι φαίνεται. Ο ιό αυτό δεν προκάλεσε τόσο μεγάλη πανδημία όσο αρχικά υποθέσαμε. Και η στάση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ε, η στάση του ήταν αρκετά αμφιλεγόμενη. Δεν πήρε θέση στο θέμα αυτό. Ολοκληρώσατε τον χρόνο σας. Η κυρία Ζαβόρσκα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρίβαζη για την περιεκτική πλήρη έκθεση. Αναφέρει ποια είναι τα σημεία για τον τομέα τη υγεία, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο επίπεδο. Η έκθεση παρουσιάζει ένα εκτενή κατάλογο μέτρων που πρέπει να αναλυθούν ώστε η κατάσταση που συνέβη το 2009 και 2010 να μην επαναληφθεί. Και όταν η πανδημία είχε προναγγελθεί, όταν προναγγέλλεται μια τέτοια σκανδαλώδε ναι. σκανδαλώδες ήταν ότι κράτη-μέλη όπω και η Σλοβακία εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ δαπάνησαν ε, για να προστατευτούν οι πολίτε έναντι μια μη υπάρχουσα απειλής. Ενδιαφέρον είναι να ξέρουμε ποιο αποκόμισε ωφέλη και επίση ποιο είναι υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση. Αυτό που αποουσιάζει από αυτή την έκθεση είναι ένα πράγμα. Η πρόταση να εισαχθεί ένα στοιχείο, ένα παράγοντα προσωπική ευθύνη υπευθυνότητα βλέπουμε ότι πιο, με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι η πανδημία επεκτείνεται αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέσλουντ θα λάβει τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπήρξε μεγάλη σύγχυση όσον αφορά τις διαφορετικές συστάσεις που προήρχονται από διαφορετικές, για διαφορετικές χώρες στην ε, δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την ε, Δημόσια Υγεία είχαμε και υπουργό από πλευρά της Σουηδίας που είχε τότε την Προεδρία στο Συμβούλιο και που είχε αναλάβει την παρακολούθηση αυτού του θέματος και ταυτόχρονα την ίδια ημέρα ε, ακούσαμε την ECDC που έδωσε τελείω άλλη αξιολόγηση τη κατάσταση και τελείω διαφορετικέ συστάσει. Ο ένα έλεγε είναι επικίνδυνη η κατάσταση, οι άλλοι έλεγαν όχι. Ήταν μεγάλη σύγχυση που είχε δημιουργηθεί και είναι δύσκολο, ήταν δύσκολο για ε, να, να μπορέσει κανεί να συναγάγει τα σωστά συμπεράσματα. Τίθεται το ερώτημα πώ πραγματικά στην πραγματικότητα θα αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα. Υπήρχε μεγάλη ζήτηση για τέτοια εμβόλια και οδηγηθήκε η κατάσταση σε χαοτική κατάσταση. Είχαν, είχαμε προβλήματα με τις αποθήκες και είχαμε διαφορετικές καταστάσεις. Ολοκληρώσατε τον χρόνο σας η κυρία Ρόιτοβα, λέγει ο Πρόεδρος. Η κυρία Ρόιτοβα, παρακαλώ, έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Τώρα εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε ότι τα δισεκατομμύρια ευρώ που επενδύσαμε για την γρήπη αυτή ήταν υπερβολικά ποσά. Αλλά ως απόφαση πρέπει να δούμε τι έκανε η Πολωνία. Δεν υπέκυψε στις πιέσεις και δεν σημειώθηκαν περισσότερα κρούσματα από ό,τι ε, αλλού που είχαν γίνει εμβολιασμοί. Ευχαριστώ λοιπόν για την έκθεση αυτή και πιστεύω ότι όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και χώρες πρέπει να πάρουν μαθήματα από την κατάσταση αυτή πρέπει οι αγιονομικές αξιολογήσεις να γίνονται σωστά ως προς τον κίνδυνο. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε. Η κυρία Εστρέλα θα λάβει τώρα τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ ήδη αναφέρθηκαν αμφιβολίες σε σχέση με τα εμβόλια για την γρήπη ή τα Και είναι φυσικό ότι οι πολίτες διαρωτώνται και έχουν κάποιες υποψίες εφόσον ήδη το 2009 υπήρξε μια εκστρατεία ενημέρωσης σε όλα τα κράτη-μέλη και έγιναν μεγάλες έρευνες και επενδύσεις, επενδύσεις όσον αφορά τα εμβόλια και ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας ανήγγειλε μια πανδημία, προανήγγειλε μια πανδημία και η κατάσταση άλλαξε άρδιν στη συνέχεια. Δηλαδή, στη συνέχεια το 2010 ουσιαστικά δεν, δεν γινόταν πλέον λόγος για την γρήπη ή τα ένα Και γι' αυτό είναι φυσικό οι πολίτες να διαρωτώνται περί τίνος πρόκειται. Αν υπήρξε κάποιος, κάποια επικινδυνότητα ή όχι τότε και τώρα. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κυρία Εστρέλα, εξαντλήθηκε ο χρόνος σας. Τώρα η κυρία Κάντενμπαχ και τωρα προεδρο σας ευχαριστω κυρια εστρελα εξαντληθηκε ο χρονος σας τωρα η κυρια καντενμπαχ και ετσι θα ολοκληρώσουμε αυτόν τον γύρο παρεμβάσεων. Παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, νομίζω ότι σήμερα πρέπει να θεωρούμε ότι είμαστε ευτυχεί ότι η πανδημία, η επιδημία δεν πήρε την εξέλιξη που είχε προαναγγελθεί. Δηλαδή σε σχέση με ε, τα πολλά θύματα που είχαν προβλεφθεί. Αλλά κάθε θάνατο είναι τραγικό γεγονό. Θέλω να πω εδώ ότι η σαφή αντανάκταση τη κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τελείω ε, διαφορετικά βιώματα από τα κράτη-μέλη. Έχουμε διαφορετικά συστήματα υγεία, διαφορετικέ δομέ. Ε, η προστασία υγεία ε, είναι εθνική υπόθεση σε σχέση με μια πανδημία. Χρειάζεται όμω η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είδαμε ότι και στα δύο επίπεδα πρέπει πολλά να μάθουμε, γιατί πολλά πρέπει να γίνουν καλύτερα. Πολλέ φορέ συζητήθηκε και το αναφέραμε σήμερα έχουμε μια κατάσταση όπου η εμπιστοσύνη των πολιτών πρέπει να ξανακερδιθεί. Η αντιμετώπιση της γρήπης ή τα 1 κατέδειξε ότι υπήρξαν ελλείψεις εδώ και ελαττώματα και πρέπει να έχουμε καλύτερο συντονισμό στο μέλλον. Σας ευχαριστώ κυρία. Ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο στην ημερησία διάταξη, λέγει ο Πρόεδρος. Κλείνουμε τη συζήτηση με την παρέμβαση της Επιτρόπου κυρίας Δαμανάκη. Παρακαλώ κυρία Δαμανάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγητρία, την κυρία Ριβαζή, για αυτή την έκθεση. Η έκθεση αυτή πραγματικά είναι μια αξιόλογη συνεισφορά στην όλη μα προσπάθεια να αντλήσουμε διδάγματα από την πανδημία του 2010. Συμφωνώ μαζί σα ότι πρέπει να μάθουμε πολλά από αυτή την εμπειρία. Και επίση πρέπει με κριτικό μάτι να δούμε πώς ανταποκριθήκαμε στην κατάσταση αυτή. Πρέπει να διασφαλίσουμε την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών έναντι τέτοιων υγειονομικών απειλών. Για αυτόν τον σκοπό πρέπει να βελτιώσουμε την ετοιμότητά μας και το σχεδιασμό μας, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες διασυνοριακές απειλές για την υγεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη είχε αυτόνομες δυνατότητες και εμπειρογνωμοσύνη για την πανδημία της γρήπης. Στον τομέα της έρευνας και μόνον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από 15 προγράμματα από το 2000 και με επενδύσεις 150 χιλιάδων τουλάχιστον ευρώ, το εκατομμυρίων ευρώ, 150 εκατομμυρίων ευρώ. Το ε, ερευνητικό μας κέντρο για την παρακολούθηση των πανδημιών ε, προ... Ε, μας έδωσε επιστημονικές συμβουλές κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής και προς τα κάτι μελη και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι, Ευρωπαϊ... οι δομές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στήριξαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας τα εθνικά κράτη στις προσπάθειές τους. Ωστόσο, όπως φαίνεται από την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, η αποτίμηση της απόκρισής μας έδειξε μια σειρά από και ε, κενά τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν. Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι προμήθεια εμβόλια για την πανδημία, η ανάγκη συντονισμού των στατηγικών εμβολιασμού, η ανάγκη ευελιξίας στα προγράμματα ετοιμότητάς μας και η ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας. Ε, εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη στήριξη ε, των επιστημονικών φορέων και με τη βοήθεια των κρατών μελών, διότι εδώ μιλάμε για κοινή αρμοδιότητα με τα κράτη-μέλη, να τελέσει πρόοδο στα θέματα αυτά. Εδώ έχουμε δύο πρωτοβουλίες τουλάχιστον. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια πρωτοβουλία για την ασφάλεια και την υγεία πριν το τέλος της χρονιάς ώστε να ενισχύσει τις δυνατότητες συντονισμού μας. Και κατά δεύτερον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανακινήσει έναν κοινό μηχανισμό ε, διαγωνισμό για τα αντιϊκά και τα εμβόλια για όσα κρατημέλη θέλουν να συμμετάσχουν σε τέτοιες διαδικασίες. Εδώ θα ενισχύσουμε την αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζοντας ένα ελάχιστο επίπεδο ισότιμης πρόσβασης σε εμβολιασμό. Και έτσι θα έχουμε και μεγαλύτερη δυνατότητα να προσπάσουμε καλύτερους συμβατικούς όρους, συμβασιακούς όρους. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τη χαρά τη για τη στήριξη της ε, εισηγήτριας για τέτοιε πρωτοβουλίε. Επίση, σκοπεύουμε να χρηματοδοτήσουμε περαιτέρω έρευνα για να δούμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά και τις αδικές επικοινωνία των ε, κρατών μελών και να βελτιώσουμε τι ε, τα προγράμματα εμβολιασμού. Επίση, περισσότερη διαφάνεια και ζητήματα ανεξαρτησία ανέκλειψαν στην έκθεση. Τα θεωρούμε πολύ σημαντικά και αυτά. Και εδώ πιστεύουμε ότι πραγματικά κάτι πρέπει να γίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρμόδιοι φορεί θα συνεργαστούν προκειμένου να βελτιώσουν τις διαδικασίες που ήδη υπάρχουν για την δήλωση συμφερόντων και την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να προκύψει. Εδώ λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε να ε, καταβάλουμε όλοι προσπάθειες προς τον κοινό στόχο ε, τη καλύτερη προετοιμασία για την προστασία των ε, συμπολιτών μα για τις μελλοντικές υγειονομικές απειλές. Σα ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Με την παρέμβαση τη κυρία Δαμανάκη ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξή μα και η ψήφιση της, ε, των αντίστοιχων προτάσεων ψηφίσματος θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη.